Καλησπέρα, συνάδελφοι. Συγγνώμη για τη μικρή καθυστέρηση. Έγκριση ημερήσια διάταξη. Σημείο 1. Έχουμε αλλάξει λίγο την ημερήσια διάταξη. Έγκριση συστάσεων των συντονιστών, όπω έχουμε στο σημείο τη 29 Ιανουαρίου των συντονιστών. Στο σημείο 2 θα το συζητήσουμε αυτό σύμφωνα με το 205 το άρθρο, στην αρχή ψηφορία τη Λίμπε στι 16 και 35 θα το συζητήσουμε. Η Σιάρα, κύριε Ντόλτον. Ευχαριστώ. Μιλώ βάσει του άρθρου 205 να ψηφίσουμε σήμερα στην Επιτροπή Λίμπε την απόφαση των συντονιστών να συντάξουμε μια έκθεση του άρθρου 7, ενδιάμεση έκθεση για την Πολωνία. Καλώς. Αν ζητά μια ομάδα σύμφωνα με το άρθρο 205 θα ψηφίσουμε. Ονομαστική θα γίνει στις 16.35 για το σημείο 4.3 του σημειώματος των συντονιστών, θέμα των πρασίνων, ψηφίστηκε με πλειοψηφία για την απόφαση για την Πολωνία. Ονομαστική ψηφοφορία 16 και 35. Σημείο 10 ψηφοφορία για την Ευρωπαϊκή Ακτοφυλακή και Μεθοριοφυλακή αναβάλλεται για 11η Φεβρουαρίου. Αυτέ είναι οι μόνε αλλαγέ. Αν υπάρχουν αντιρρήσει, εγκρίνεται τροποποιηθήσα ημερήσια διάταξη. Καλώ. Πάμε λοιπόν στις ανακοινώσει. Έχουμε διερμηνία σε όλε, τις γλώσσες από δανέζικα, γοδελικά και κροατικά. Και έχουμε έγκριση συστάσεων των συντονιστών άρθρο 205 κλπ. λοιπά Και κάποιες πληροφορίες για εφαρμοστικές πράξεις και καταξιοσυδότηση πράξης. Αν θέλει κάποιος να υποβάλει ενστάσεις, πρέπει να ενημερώσει δόντως την γραμματεία της ΛΥΜΠΕ πριν την 11η Φεβρουαρίου 12 μεσημέρι. Πάμε στο σημείο 3. διάδοση τρομοκρατικού περιεχομένου στο διαδίκτυο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο Κοινοβούλιο υπέβαλε πρόταση για την πρόληψη τη διάδοση περιεχομένου τρομοκρατικού στο διαδίκτυο το φθινόπωρο πέρασε. Η πρόταση είναι άλλο ένα βήμα σε σειρά μέτρων και πρωτοβουλειών που έχουν σκοπό να εξασφαλίσουν το ότι το διαδίκτυο χρησιμοποιείται για τη διάδοση τη τρομοκρατία και τρομοκρατική προπαγάνδα και τρομοκρατικού περιεχομένου πρέπει να αφαιρείται γρήγορα. Και αυτό το θέμα είναι πάρα πολύ ευαίσθητο και σημαντικό, αυτό είναι προφανές και είναι πολύ σημαντικό για το έργο της Επιτροπής μας. Όμως οι συζητήσεις της προτάσεως καθυστέρησαν λόγω συγκρούσεως αρμοδιοτήτων και συζητήσεων ΙΜΚΟ και ΚΟΥΛΤ και τώρα επελήθη το πρόβλημα και έχουμε διευθέτηση μεταξύ των δύο επιτροπών. Ο εισηγητής θα τα εξηγήσει σίγουρα αυτά. Συνάδελφοι, νομοθετικοί φάκελοι, προτεραιότητες, ένα για την, είναι για την υπόλοιπη θητεία και προσδοκίες που έχουμε είναι ότι η Επιτροπή ΛΥΜΠΕ θα μπορέσει γρήγορα να εγκρίνει την έκθεσή της χωρίς να χρονοτριβήσω. Θα δώσω το λόγο στον εισηγητή για να παρουσιάσει το σχέδιο έκθεσης. Ο Dan Dalton, λοιπόν που είναι εισηγητής μπορεί να παρουσιάσει το θέμα. Νταν, ευχαριστώ Πρόεδρε. Να αναφέρω ποια είναι η κατάσταση των φορά της μακρές οι συζητήσεις. Και αυτό μας περιέπλεξε σε εργασίες. Η Επιτροπή ΙΜΚΟ έχει αρμοδιότητα για τα ενεργά μέτρα μαζί με μας. Παρόλο που εμείς ελέγχουμε αυτό το θέμα, η Επιτροπή Πολιτισμού έχει αρμοδιότητα για τα οπτικοακουστικά Τα οπτικοακουστικά καλύπτουν την τρομοκρατία στο διαδίκτυο μεγάλο κομμάτι του θέματο. Άρα πρέπει να συνεργαστούμε στενά και με τι δύο επιτροπέ, αλλά κυρίω με την Επιτροπή Πολιτισμού. Και αυτό περιπλέκει το χρονοδιάγραμμα κατά κάποιο τρόπο. Όμω, στόχο μου είναι να εξασφαλίσω ότι τουλάχιστον θα έχουμε θέσει το Κοινοβουλίο ετοίμητο διαπραγμάτευση με το Συμβούλιο πριν το τέλο τη θητεία. Το Συμβούλιο θέτησε τη θέση του το Δεκέμβριο και υπάρχουν πολλέ προσδοκίε ότι γρήγορα θα διεκπαιρεωθεί το θέμα Άρα δεν νομίζω ότι ως Κοινοβούλιο και σαν Επιτροπή θέλουμε να δώσουμε την εντύπωση ότι εμείς καθυστερούμε και κολλησιεργούμε όσον αφορά τη θέση μας. Υπάρχει σαφώς ανάγκη για το νομοθέτημα αυτό. Η ριζοσπαστικοποίηση στο διαδίκτυο είναι βασικό στοιχείο της ριζοσπαστικοποίησης ανθρώπων και οι περισσότεροι δέχονται ότι οι πλατφόρμες που να κάνουν πολλά περισσότερα σε σας εξασφαλίσουν αυτό το περιεχόμενο δεν θα είναι διαθέσιμο στις πλατφόρμες τους. Νομίζω ότι είναι σαφές ότι όλοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση προς εμάς προσβλέπουν για να το καταφέρουμε αυτό. Τώρα γενικά, σαν αποτέλεσμα των εργασιών, στόχος της προτάσης μπορώ να πω ότι είναι σωστός, πρέπει όμως να έχει καλύτερη στοχοθέτηση για να είναι αποτελεσματική η προσέγγιση και αυτό αφορά ιδιαίτερα την ελευθερία της έκφρασης και της ενημέρωσης και προσπάθησα αυτό το πετύχω στη ώστε Θα διατρέξω εντάχει τους βασικούς ε, τομεί που, δημιουργεί, που δημιουργούν ησυχίε. Το πεδίο εφαρμογή. Όσον αφορά το πεδίο εφαρμογή τη προτάσεω, πρέπει να δούμε πόσο πρέπει να εφαρμόζεται στις μικρομεσαίες επιχειρήσει, σε ποιο βαθμό θα πρέπει να εστιάζεται επί στο σελίδων υψηλού κινδύνου. Όμως προσωπικά δεν θέλω να προβλέψω γενικούς, ε, γενικές εξαιρέσεις και όρια που αυτό δείχνει ότι έχει αποτύχει νομοθεσία. Πρέπει να γνωρίσουμε ότι οι μικροσυρέ επιχειρήσει σε αυτή την περίπτωση πολύ συχνά είναι οι πλατφόρμε που απειλούνται περισσότερο από αυτό το περιεχόμενο. Και ε, στην προσπάθειά του να βγάλουν το περιεχόμενο από τι ιστοσελίδε του. Πρέπει να προσέξουμε την προσέγγιση μα. Εν γέννη, λοιπόν, το πεδίο εφαρμογή μεταλογικό Δεν νομίζω ότι η υποδομή για τι υπηρεσίε ε, ε τι είναι κάτι καλό. Δεν μιλάει για Dropbox, αλλά υποδομέ νεφοϋπολογιστικές που χρησιμοποιούνται από επιχειρήσεις για αποθήκευση στοιχείων. Δεν έχουν τα στοιχεία αυτά και δεν μπορούν να αφαιρέσουν συγκεκριμένο περιεχόμενο. Πρέπει να κατεβάσουν ολόκληρε σελίδε για να πετύχουν ένα συγκεκριμένο κομμάτι τρομοκρατικό σε συγκεκριμένη σελίδα. Οπότε αυτό δημιουργεί και δεντολογικό πρόβλημα. Διότι η πλατφόρμα διαδίδει τι πληροφορίε προ του καταναλωτέ και όχι η εταιρεία που ε, Έχετε στο σελίδα. Η πλατφόρμα είναι που διαδίδει το περιεχόμενο και θα πρέπει να είναι το, ο πρώτος στόχος των αρμοδίων αρχών και τα μέτρα ε, θα πρέπει σε αυτούς να εφαρμοστούν αν δεν συμμορφωθούν. Πολλοί άλλοι ορισμοί της προτάσεως ήδη έχουν τυποποιηθεί στην νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, αλλά το πιο προβληματικό θέμα είναι ο ορισμός του τρομοκρατικού περιεχομένου, αυτός καθεαυτός. Κατά την άποψή μου, ο καλύτερος τρόπος να αντιμετωπιστεί είναι να ο ορισμός με την οδηγία τρομοκρατίας που περιέχει ήδη ορισμό, ξέρω ότι είναι ατελής, αλλά είναι ότι καλύτερο έχουμε στη διάθεσή μας. Και δεν νομίζω ότι θα πρέπει σε αυτή τη φάση να ανοίξουμε αυτό το θέμα και να αρχίσουμε τώρα συζήτηση τι πρέπει να θεωρηθεί σαν τρομοκρατικό περιεχόμενο και τι όχι. Αλλιώ βρισκόμαστε τη θέση όσον αφορά τις διάφορες πολιτικές απόψεις που επικρατούν στον κόσμο. Οπότε είναι καλύτερο πραγματικά να ευθυγραμμιστούμε με τον ορισμό περί τρομοκρατίας, τρομοκρατικού περιεχομένου στην οδηγία περί τρομοκρατίας. Επίσης δύσκολο σχετικά με αυτό οι πλατφόρμες να καθορίσουν ποιο περιεχόμενο παράνομο και όποιο όχι. Οι επιχειρήσεις δεν πρέπει να βρεθούν σε αυτή τη θέση που θα πρέπει να κρίνουν, διότι αν βρεθούν σε αυτή τη θέση ιδιωτικά θα θέσουν μεγαλύτερα, πιο αυστηρά όρια όσον αφορά τη λογοκρισία από ό,τι θα έπρεπε. Είναι σαφέ ότι οι αρχές θα πρέπει να παράσχουν ακριβεί κατευθύνσει επ' αυτού και δεν θα πρέπει αυτό να το αφήσουμε στι σελίδε να αποφασίσουν. Διότι εκεί ελοχεύει ο μεγαλύτερο κίνδυνος για τα θεμελιώδη δικαιώματα. Μεγάλη ανησυχία στην πρόταση είναι κάτι άλλο η διατάξη περισμένων ευθυνών στην οδηγία περί ηλεκτρονικού εμπορίου στου δικαιού και η διατάξη του κανονισμού επιτρέπουν στα κράτη-μέλη να επιβάλλουν ενεργώ μέτρα στου παρόχου υπηρεσιών που φιλοξενούν τι σελίδε. Θα πρέπει να φύγουν την κατάσταση όπου η υποχρέωση για γενική παρακολούθηση επιβάλλεται από την πίσω πόρτα μέσω του κανονισμού. Έκανα αλλαγέ στο άρθρο 6 προσπαθώντα να περιορίσω την εθελοντική επιβολή ενεργών μέτρων σε περιπτώσει όπου ε, όπου έχουν δοθεί, εκδοθεί πολλές εντολές αφαίρεσης α, ε, περιεχομένου σε ιστοσελίδα. Αυτή η ιστοσελίδα δηλαδή είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη. Αν αυτό το όριο το προσέξουμε θα σβήσουμε σχεδόν όλες τις ιστοσελίδες και τα μέτρα θα πρέπει να εφαρμοστούν σε στοχευμένα. Δεν θα υπάρχει γενικός έλεγχος και παρακολούθηση. Και τα θελοντικά μέτρα που λαμβάνονται από τι πλατφόρμε θα πρέπει να λαμβάνονται πλήρω υπόψη όταν εξετάζουμε κατά πόσο συμμορφώνονται με τον κανονισμό οι πλατφόρμε. Ξέρω ότι υπάρχουν όμω πολλέ ανησυχίε για το Κοινοβούλιο για παραβιάσει τη ελευθερία του λόγου, δυνάμει το άρθρο 6, και με τα χαρά συνεργαστώ στενά με συναδέλφου ε, για να βρούμε άλλε λύσει στο μέλλον. Δεν πιστεύω όμω ότι η διαγραφή πλήρη του άρθρου είναι η καλύτερη προσέγγιση. Κάποια μέτρα θα μπορούσαν να έχουν θετικότατο αντίκτυπο όσον αφορά την αντιμετώπιση του δημοκρατικού περιεχομένου, αλλά μόνο οι πλατφόρμε αυτέ οι οποίε δημιουργούν τον κίνδυνο και έχουν αρνηθεί να συνεργαστούν με τι αρχέ. Στον κανόνα περί αυτό είναι βασικότατο σημείο της προτάσεως, ε, επίμαχο θέμα, κανόνος για ε, όριο μια ώρα για την αφαίρεση κατόπιν εντολή. Οι αρχέ επιβολή του νόμου κατέστησαν σαφέστατο σε μένα πόσο ζωτική είναι η αρχή τη μία ώρα για να αποφυγεί να αποφύγουμε τη διάδοση την ταχεία του περιεχομένου. Στην πρώτη ώρα λοιπόν το περιεχόμενο αυτό διαδίδεται στο μέγιστο βαθμό. Εγώ έθεσα πολλέ ερωτήσει. Του είπα μέχρι έρθει να έρθει μια εντολή, το περιεχόμενο ήδη είναι πάνω από μια ώρα στο διαδίκτυο. Αν η πρώτη ώρα είναι η δικαιολόγηση για την προθεσμία τη μια ώρα, θα πρέπει να το εξετάσουμε ξανά το θέμα, διότι είναι σαφέ πόσο έχει ανέβει αυτό το περιεχόμενο πριν εκδοθεί εντολή. Και αυτή είναι η ερώτηση που έχουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και του άλλου εμπειρογνώμονε. Το περιεχόμενο πόση ώρα είναι στην σελίδα πριν το πάρουν χαμπάρι. Έτσι αυτό επηρεάζει και πώ θα συζητήσουμε το θέμα τη μια ώρα. Αυτό το κείμενο έχει στην πρότασή μου. Όμως με διάφορα μέτρα χαλαρωτικά. Θα πρέπει να υπάρχει επικοινωνία πρώτα απ' όλα μεταξύ αρμόδιας αρχής και πλατφόρμας πρώτα και θα πρέπει να ξεκινήσει η εντολή εκτός εντολής αν αρνηθεί η πλατφόρμα να συμμορφωθεί, να βοηθήσει να επικοινωνήσει με τις αρμόδιες αρχές. Πιστεύω ότι αυτό περιορίζει τον αντίκτυπο του μέτρου της μίας ώρας κατά κάποιο τρόπο. Όμως υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με την μία ώρα τεράστιες πλατφόρμες θα έχουν τα μέσα να κατεβάσουν το περιεχόμενο σε μία ώρα. Πιθανότατα, συνήθως, αλλά για μικρή πλατφόρμα, μία-δύο τέτοιε πολύ μικρέ πλατφόρμε, αυτό θα είναι δυσχερέστατο. Οι μικρομεσαίε επιχειρήσει σίγουρα μπορεί να μην τηρήσουν μια προθεσμία, κυρίω αν είναι στη διαφορετική ζώνη χρονική. Οπότε θα πρέπει να το επεξεργαστούμε αυτό το θέμα τη μια ώρα και είμαι ανοιχτό. Μπορώ να συνεργαστώ με του κοιόδη για να βρούμε κάτι το οποίο θα λειτουργεί οι μικρότερες ιστοσελίδες που ανέφερα έχουν και μικρότερο ακροατήριο, οπότε κανονικά ο κίνδυνος που δημιουργούν είναι μικρότερος για διάδοση τρομοκρατικού περιεχομένου, αλλά όχι πάντα βέβαια. Πολύ συχνά μια μικρή ιστοσελίδα που μπορεί να έχει πολλές συγκεκριμένους ε, θεατέ με παρόμοιε απόψει, παρόλο που είναι πολύ μικρή ιστοσελίδα, μπορεί να παίξει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο στη ρίζοσπαστικοποίηση. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να είμαστε κάπω προσεκτικοί Ποιου θα εξαιρέσουμε αν εξαιρέσουμε τι μικρομεσαίε επιχείρησει. Επίσης προτείνω να περιορίσουμε τις αρμόδιες αρχές που μπορούν να εκδώσουν αυτή την εντολή αφαίρεσης να είναι μια αρχή σε κάθε κάτω μέλος εκτός αν οι συνταγματικές διευθετήσεις το καθιστούν αυτό ανέφικτο. Αν περιορίσουν τον αριθμό των αρχών αυτών, θα μπορούν οι πάροχοι υπηρεσιών να είναι πεπισμένοι ότι δέχονται μια εντολή που είναι πραγματική και να μην έχουμε υπερβολικό άχθο αλληλεπικάλυψη, εάν υπάρχουν πολλέ αρχέ που παρεμβαίνουν. Προτείνω και ένα άρθρο 15 που απευθύνει δυνατότητα έφεσης. Ε, η εταιρεία μπορεί να υποβάλει έφεση στην νομική, στη χώρα στην οποία έχουν νομική εκπροσώπηση. Σχετικά με αυτό είναι σημαντικό, δυνάμει το άρθρο 8, να απαιτείται η αρμόδια αρχή να δημοσιεύει εκθέσει διαφάνεια περί δράσεω που έχει αναλυφθεί κατά τρομοκρατικού περιεχομένου, κυρίω να αναφέρονται σε περιπτώσει το περιεχόμενο λανθασμένο εντοπίστηκε στο τρομοκρατικό. Ανθρώπινη υποπτία δύσκολων υποθέσεων είναι κρίσιμη σημασία και ενίσχυσε αυτή την απέτηση στο άρθρο 10. Παρόμοιε καταγγελίε για άρση του περιεχομένου πρέπει γρήγορα να εξετάζονται από του παρόχου, γι' αυτό βάλαμε και δύο εβδομάδε σαν προθεσμία. Τώρα, κυρώσει. Σημαντικό κομμάτι ε, τη προτάσεως θέλουμε ευέλικτο σύστημα κυρώσεων που αναγνωρίζει ε, διάφορα ελαφρυντικά, κυρίω όταν μιλάμε για 4% κύκλο εργασιών βάσει ε, τη εντολή που δίνεται για αφαίρεση εντό μια ώρα. Οπότε πρέπει να λάβουμε υπόψη και πόσο δουλεύει αυτή η ιστοσελίδα πριν επιβάλλουμε κυρώσει. Οι κυρώσει θα πρέπει να επιβάλλονται άμα συστηματικά δεν συμμορφώνται με τον κανονισμό και οι περιορισμένε δυνατότητε που έχουν οι μικρομεσαίε επιχειρήσει πρέπει να είναι ελαφρυντικό. Χωρί δίκαιη και λογική διαδικασία θα προσπαθούν να αυτοπροστατευτούν οι επιχειρήσει και θα υπάρχει μεγαλύτερη λογοκρισία ή θα προσπαθήσουν να αποφύγουν την επιβολή κυρώσεων. Κλείνοντα, πιστεύω ότι χρειάζεται αυτή η νομοθεσία, αλλά πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι αυτή η νομοθεσία αποφεύγει η νομοθεσια αποφευγει λογοκρισία η υπερβολική λογοκρισία τη τι αρχέ θα πρέπει είναι ένα σαφέστατο ορισμό τη τρομοκρατία, να μην υπάρχουν αμφισβητήσει, να είμαστε σίγουροι κατά την απόψή μα δεν υπάρχει γενική υποχρέωση ελέγχου, να μην υπονομεύσουμε την οδηγία του ηλεκτρονικού εμπορίου, του το τρόπο, αλλά θα πρέπει να έχουμε κάτι το οποίο να δώσει στι αρμόδιε αρχέ κάποια δύναμη να αντιμετωπίσουν το θέμα. Αυτά τα εισαγωγικά μου σχόλια προσβλέπω στο να ακούσω τις ε, απόψεις των συναδέλφων από αυτό. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Οι σκιώδεις τι έχουν να πούν. για το ΕΛΚ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμοι συνάδελφοι, να ευχαριστώ πρώτα απ' όλα τον εισηγητή, τον κύριο Ντάλτον, για αυτήν την κρίσιμη ε, έκθεση ε, την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Είναι λίγος ο χρόνος που έχουμε μέχρι το τέλος της θητείας. Είναι απαραίτητο λοιπόν σήμερα να προχωρήσουμε με το κείμενο αυτό. Συμφωνώ και στηρίζω απόλυτα τον εισηγητή σε ό,τι αφορά το χρονοδιάγραμμα, να εγκριθεί δηλαδή το κείμενο αυτό πριν τελειώσει η θητεία μας. Αυτό είναι αδιαπραγμάτευτο. Το διαδίκτυο είναι ο αδύναμος κρίκος ε, στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας και της ριζοσπαστικοποίησης. Ε, όλες οι τραγικές ε, τρομοκρατικέ επιθέσεις το αποδεικνύουν δεν μπορεί ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση να θεωρηθεί υπεύθυνο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να θεωρηθεί υπεύθυνο για τι καθυστερήσει στην ψήφιση ενό μια κρίσιμη νομοθεσία για την ασφάλεια των Ευρωπαίων. Βεβαίω, ε, οι γίγαντε του διαδικτύου έχουν καταργήσει το περιεχόμενο, το τρομοκρατικό περιεχομένο στι πλατφόρμε, αλλά αυτό δεν αρκεί. Το σύνολο ψηφιακών πλατφόρμων πρέπει να ασχοληθεί με το θέμα αυτό και πρέπει να τι υποχρεώσουμε και να τι βοηθήσουμε να αναλάβουν δράση. Αυτό είναι και το νόημα αυτή τη νομοθεσία. Η πρόταση λοιπόν τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι μια καλή βάση εργασία. Με ένα τέτοιο κανονισμό, ο στόχο είναι να προστατεύσουμε του Ευρωπαίου πολίτε. Αντιμετωπίζουμε εδώ κάποιε ε, οργανώσει ε, βάρβαρε οι οποίε ε, αυτή τη στιγμή καταστρέφουν την νεολαία μα. Βεβαίω, κάποιε πλατφόρμε αντιμετωπίζουν δυσκολίε στο να προσαρμοστούν, αλλά δεν μπορούμε από την πλευρά μα να δεχτούμε καμία χαλάρωση και όταν θερήσαμε να δημιουργήσουμε αυτήν την ποινική ευθύνη των μεγάλων εταιριών στο διαδίκτυο, μα είπαν ότι δεν γίνεται. Τελικά όμω, όταν εγκρίθηκε η νομοθεσία, μπόρεσαν να αφαιρέσουν περιεχόμενο. Πρέπει λοιπόν να συνεργαστούμε, να βρούμε λύσει και να στείλουμε ένα μήνυμα ε, σταθερό για το ζήτημα αυτό. Θα πρέπει επίσης όλες οι επιχειρήσεις να συμμετέχουν σε αυτή την καταπολέμηση της ψηφιακής ε, τρομοκρατίας αναπτύσσοντας τα κατάλληλα εργαλεία για να εντοπίζουν και να αφαιρούν παράνομο περιεχόμενο. Η αντίθεση σε, μια, ένα τόσο ε, ευαίσθητο ζήτημα δεν έχει νόημα και αντιπαράθεση. Είμαι βέβαιο ότι με του κοιότητε μπορούμε να βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο το κείμενο, να επιφέρουμε τι απαραίτητε διευκρινήσει, έτσι ώστε το κείμενο αυτό να αποτελέσει ένα πραγματικά χρήσιμο εργαλείο που να μπορεί να εφαρμοστεί χωρί αμφισημίε όσο γίνεται πιο γρήγορα. Αγαπητοί συνάδελφοι, ε, επιμένω ότι είναι θέμα πολιτική βούληση. Είμαστε πολιτικοί ηθήνοντε, εμεί είμαστε αυτοί που θα πρέπει να το κάνουμε να προχωρήσει. Ε, είναι για λόγους τιμή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι, γίνεται αυτό στο όνομα των, πολι, των συμπολιτών που τους οποίου εκπροσωπούμε δεν μπορούμε αυτό να το καταλήψουμε επειδή τελειώνει η θητεία μας. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ. Να ακούσουμε τώρα τον κύριο Βάιντεν Χόλτσερ από τους Σοσιαλδημοκράτες. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε να ευχαριστήσω τον εισηγητή. Προσπάθησα να λάβω υπόψη τι διάφορε αντιρρήσει που ήρθαν και εκτό ε, από τα έξω ε, για την έκθεση για να έχουμε μια λογική βάση. Το μεγάλο πρόβλημα το οποίο έχουμε είναι η πίεση του χρόνου πληροφορήθηκα ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί ε, όταν ασκούμε χρονική πίεση αλλά έχω μάθει επίσης όταν έχει νόημα να γίνεται κάτι τέτοιο πέρα δηλαδή από όλη αυτήν την συζήτηση ε, γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να έχουμε και μια έντονη συζήτηση με τον εισηγητή. Για την δική μου την ομάδα θα ήθελα να πω ότι χρειάζεται νομίζω περισσότερη ε, συνεννόηση και κάποιες περισσότερες ε, πληροφορίες τώρα. Επί της αρχής υπάρχουν κάποια πράγματα που θέλουμε να τονίσουμε. Αφενός είναι ότι πρέπει να αποφευχθεί η ιδιωτική επιβολή ε, του δικαίου υπάρχει, υπάρχουν ε, δημόσιοι μηχανισμοί επίσης ε, τα αυτόματα φίλτρα όπου δεν θα αποφασίζει ο άνθρωπος αλλά οι μηχανές είναι κάτι με το οποίο έχουμε πολλά αρνητικά παραδείγματα ήδη στα κοινωνικά δίκτυα και οδηγούνται εις άτοπον καμιά φορά Επίσης ε, τα, τα ένδικα μέσα μου φαίνονται ένα σημαντικό κομμάτι αυτής της συζήτησης ε, ή τι γίνεται εκεί πέρα στην πράξη. Και τέλος, κάτι το οποίο θα ήθελα να αναφέρω και ανέφερε νομίζω αναλυτικά ο εισηγητής είναι το θέμα του κανόνα της μίας ώρας. Από αστυνομική σκοπιά είναι πολύ λογικό και ακούγεται λογικό αλλά αν το σκεφτεί κανείς έχει κάποια μειονεκτήματα. Ποιος θα το κάνει, αν είναι μεγάλος ή μικρός, αλλά και το ερώτημα πότε συμβαίνει. Υπάρχουν και διαφορετικές χρονικές ζώνες, οι άνθρωποι κοιμούνται, όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά οι τρομοκράτες δεν κοιμούνται. Κοινούνται κινούνται 24 ώρες το 24ωρο. Οπότε υπάρχει μια ενδιαφέρουσα συζήτηση. Έχουμε κάποιες ε, επιφυλάξεις αρχής, αλλά είναι σημαντικό αυτά τα πράγματα να ξεκαθαρίσουν και να κάνουμε μετά το επόμενο ε, βήμα. με την απαραίτητη πάντα επιμέλεια και είμαι σίγουρος ότι ο εισηγητής εδώ πέρα είναι διατεθειμένος να κάνει κάτι τέτοιο. Και για την Άλντε η Μάιτε. Ευχαριστώ πολύ. Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τον εισηγητή που έκανε μια προσπάθεια Εξηγώντα προ τα πού μπορούμε να κινηθούμε, διευκρινίζοντας ε, τις αμφιβολίες που μπορουμε να κινηθουμε διευκρινιζοντας τις αμφιβολιε που υπηρχαν στο σχέδιο αυτό και είμαστε στη διάθεσή του για να εντατικοποιήσουμε τι εργασίε μας μιας και έχουμε λίγο χρόνο. Εάν θέλουμε λοιπόν να προσπαθήσουμε να ολοκληρώσουμε αυτή την προσπάθεια θα πρέπει να εργαστούμε σκληρά διότι πρέπει να δοθούν διευκρινήσει. Υπάρχει το θέμα του πεδίου εφαρμογή, των ορισμών, τα ζητήματα νομική ασφάλεια. Όλα αυτά τα θέματα δεν είναι δευτερεύοντα. Ο διάβολο κλείβεται στι λεπτομέρειε. Και επειδή μπαίνουμε σε ένα ζήτημα που έχει να κάνει με τον, την ιδιωτική ζωή, ε, τη, δημο, το δημο, τη δημόσια ζωή, την ελευθερία έκφρασης, θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Πρέπει να είναι λεπτομερή αυτά που λέγονται όταν μιλάμε για απαιτήσει σε δημόσιο επίπεδο. Γνωρίζουμε ότι δεν είναι το ίδιο ε, αυτό που ισχύει για τις επιχειρήσεις και αυτό που ισχύει ε, για τις ανοιχτές πληροφορίες που είναι διαθέσιμες δηλαδή στο κοινό. Θα πρέπει να βασιστούμε ε, σε αυτά που μας λέει η Οδηγία για τα πολέμηση της τρομοκρατίας. Ε, ιδάλλως δεν θα προλάβουμε. Έτσι λοιπόν συμφωνούμε μαζί σας ότι ε, εκτός της που δεν γίνεται για λόγους νομοθετικούς πρέπει να υπάρχει μία μόνο αρμόδια αρχή ε, και δεν μπορεί να υπάρχει ε, λογοκρισία προς τους ιδιώτες ε, διότι αντιβαίνουμε βασικές αρχές μας. Πρέπει να είμαστε πολύ συγκεκριμένοι στο τι θέλουμε να πετύχουμε, να έχουμε ένα σύστημα όσο γίνεται πιο απλό και να επιβαρύνει αυτό όσο γίνεται λιγότερο, ιδίως στους μικρούς παρόχους. Στην τροπολογία 34 μιλάτε για μεγαλύτερη ευελιξία απέναντι στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όχι μόνο συμφωνούμε, αλλά πρέπει αυτό να το εξηγήσουμε ακόμα περισσότερο. Διότι οι δημόσιες αρχές δεν μπορούν να επιβάλλουν δυσθεώρητα ε, μέτρα σε επιχειρήσεις που δεν έχουν τα μέσα να τα εφαρμόσουν. Ε, θα πρέπει λοιπόν να δούμε και το θέμα των προθεσμιών, το θέμα των λαθών, των συστηματικών λαθών ή βεβαίω και την κακή πίστη. Έτσι. Όλα αυτά όμω πρέπει να αποδεικνύονται. Ε, γι' αυτό υπάρχει και ο έλεγχο ο δικαστικό. Εφόσον υπάρχει έλεγχο δικαστικό στον πραγματικό κόσμο, πρέπει να υπάρχει και στο ψηφιακό. Πρέπει να είμαστε λοιπόν αναλογικοί ε, στην χρήση του καθενό από αυτά τα εργαλεία. Τώρα, όπω είπατε κι εσείς, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μα ε, και του περιορισμένου ανθρώπινου πόρου των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ε, δεν ξέρω αν πρέπει να δοθεί κάποιο άλλο κίνητρο σε αυτέ τι επιχειρήσει για να μπορέσουν να εφαρμόσουν αυτά τα μέτρα, ίσως να προλεφθούν κάποια μέτρα υποστηρικτικά, ε, ανάλογα με το στόχο που θέλουμε να πετύχουμε τελικά. Τώρα, όταν μιλάτε για ενεργητικά μέτρα, στο άρθρο 6 ή στο άρθρο 8 μπορεί να υπάρχουν εδώ κάποια κάποιες ελλείψεις. Ε, εμείς ε, εδώ θέλουμε αναλογικότητα. Θέλουμε να είναι απλά τα πράγματα και να είναι εφαρμόσιμα. Ο καθένας δηλαδή να κάνει την προσπάθεια που τον αλογεί με βάση τη θέση που έχει στο σύστημα αυτό και στην κοινωνία γενικότερα. Για τις προθεσμίες μίλησα. Τα κράτη-μέλη που έχουν την ευθύνη για να καθορίσουν ότι και να κρίνουν ότι το περιεχόμενο είναι τρομοκρατικής φύσης είναι αυτά που θα πρέπει να καθορίσουν και που μπορούν να μπορούν να το καθορίσουν αυτό γρήγορα. Τα υπόλοιπα θα πρέπει να τα δούμε εμείς ε, στη συνεργασία που θα έχουμε. Και εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να έχουμε όσο γίνεται λιγότερες ε, ε, διτές επιλογές, τα άρθρα 4 και 5 με την απόσυρση ε, όσο γίνεται λιγότερες ε, λοιπόν ε, αμφίσιμες επιλογές, όσο γίνεται πιο συγκεκριμένοι να είμαστε, ο δικαστικός έλεγχος πρέπει να είναι απολύτως ρητός, πρέπει ο μηχανισμός γενικά να περιγράφεται ρητά έτσι ώστε όλοι να ξέρουν τι τους περιμένει ε, ώστε τα λάθη δηλαδή να μην οφείλουν στην αφησιμία της πρότασης να μπορούμε πραγματικά να βοηθήσουμε να είναι ελάχιστα αυτά τα λάθη και όταν βεβαίω δεν υπάρχει καλή πίστη να μπορούμε αυτό να το εντοπίσουμε. Είναι σημαντικό το ζήτημα αυτό, ξέρουμε ότι πρέπει να γίνει μια προσπάθεια να προχωρήσει, είμαστε στη διάθεσή σας, αλλά η νομική ευθύνη, η νομική ε, ε, ασφάλεια είναι πολύ σημαντική. Όλοι οι ορισμοί, οι ορισμοί, το περίφαρμογής πρέπει να είναι πολύ συγκεκριμένοι δεν μπορούμε να κατακλείσουμε τους μικρούς παρόχους υπηρεσιών, να τους πνίξουμε στους κανονισμούς και πρέπει να έχουμε κατά νου τι μπορεί, τι μπορεί να συμφορά της Επιτροπής ΙΜΚΟ και της Επιτροπής ΚΟΥΛΤ. Θα σας συνδράμουμε έτσι ώστε μέσω των τροπολογιών όλα αυτά τα ζητήματα που μας απασχολούν και βλέπω ότι είμαστε πολύ αυτοί που τα παραλαμβάνουν να μπορέσουμε να οδηγήσουμε, να οδηγήσουμε, σε, να οδηγήσουμε το κείμενο σε κάτι ε, χρήσιμο και να μην μπερδεύουμε τα πράγματα. Αναλογικότητα λοιπόν. Εφόσον υπάρχει αναλογικότητα, εμεί θα σα υποστηρίξουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και Βαζολή τώρα για τους πράσινους. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τον εισηγητή της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ αλλά και τους εισηγητές της ΚΟΥΛΤ και της ΙΜΚΟ για την πρόταση έκθεση ό,τι αφορά την απόσταση τρομοκρατικού περιεχομένου επιγραμμικά. Ε, νομίζω ότι όλοι συμμεριζόμαστε τον στόχο. Εδώ δεν υπάρχει ε, καμία αμφιβολία από αυτού. Ξέρουμε ότι η ριζοσπαστικοποίηση των διαφόρων ατόμων δεν γίνεται μόνο στο διαδίκτυο βέβαια, παρότι το διαδίκτυο συνεισφέρει σε, αυτό, σε, αυτήν, σε, σε αυτόν σημαντικά. Ε, υπάρχουν αποκλήσεις ό,τι αφορά τα μέσα, ό,τι αφορά τη μέθοδο που θα μας ε, οδηγήσει στην απόσυρση του περιεχομένου. Διότι δεν θέλουμε ένα διαδίκτυο το οποίο είναι στην υπηρεσία μιας τρομοκρατικής προπαγάνδας, αλλά δεν θέλουμε και ένα διαδίκτυο το, όπου θα υπάρχει ε, διαδεδομένη λογοκρισία και τις οποίες, το οποίο το περιεχόμενο θα, θα καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από τους μεγάλους γίγαντες τους ψηφιακούς. Δηλαδή, η καταπλέμιση της δημοκρατίας δεν μπορεί να οδηγήσει σε δυσανάλογες επιθέσεις και περιορισμούς των θεμελιών δικαιωμάτων. Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά δημοκρατικό περιεχόμενο επιγραμμικά, χωρίς να διακυβεύεται η ελευθερία έκφραση του καθένα να μην κινηθούμε δηλαδή σπασμωδικά χωρίς να σκεφτούμε τις ε, επιπτώσεις. Ας προχωρήσουμε θέλοντας τα σωστά ερωτήματα. Σε αυτό το πνεύμα λοιπόν αναλογικότητας, ε, δικαιοσύνης και αποτελεσματικότητας σκοπεύω να υποβάλω τροπολογίες στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Παραδείγματο χάρη, μία από τι εγγυήσει που θα πρέπει να ενισχύσουμε είναι η φύση των αρχών που θα είναι επιφορτισμένε με την απόφαση τη ε, απόσυρση του περιεχομένου πρέπει να είναι κατά προτεραιότητα δικαστικό αυτό το όργανο. Και αν δεν είναι δικαστικό, θα πρέπει να είναι κάποιο θεσμό που θα δίνει, θα έχει όλα τα εχέγγυα ασφάλεια και δικαιοσύνη. Θα πρέπει επίση να συμφωνήσουμε ε, γύρω από τον όρο τρομοκρατικό περιεχόμενο, έτσι ώστε να μην υπάρξει κατάχρηση. Και αυτό είναι κάτι το οποίο εμένα με ευαισθητοποιεί ιδιαίτερα, διότι στη Γαλλία έχει χρησιμοποιηθεί και στο παρελθόν η νομοθεσία κατά της τρομοκρατίας κατά πράσινων ακτιβιστών, περιβαλλοντικών ακτιβιστών, περασπιστών του περιβάλλοντος. Και όλοι ξέρουμε τι συνέβη. Ορισμένε φορέ λοιπόν, όταν υπάρχει ένα τέτοιο εργαλείο, γίνεται κακή χρήση του εργαλείου αυτού για κακό σκοπό. Τώρα, η ιδέα των υποχρεώσουμε τι πλατφόρμες να πάρουν οι ίδιε συνεργετικά μέτρα η δική μου ομάδα θεωρεί ότι αυτό δεν πρέπει να οδηγήσει de facto στην υποχρέωση της ε, θέσπισης ε, αυτοματοποιημένων φίλτρων ε, κατεβάσματος ε, περιεχομένου. αυτό οδηγεί σε περιορισμό της ελευθερίας, τα φίλτρα μπλοκάρουν υπερβολικά πολύ περιεχόμενο και υπάρχει βεβαίως και διασυνοριακή πτυχή του ζητήματος. Πιστεύουμε, θεωρούμε ότι μια δημόσια αρχή ενός κράτους μέλους να μπορεί να δώσει ε, οδηγίες σε μια επιχείρηση που βρίσκεται σε άλλη χώρα. Δεν θα ήθελα εγώ η Ουγγαρία να υποχρεώσει μια γαλλική πλατφόρμα χωρίς έλεγχο να αποσύρει κάποιο περιεχόμενο. Θα πρέπει να υπάρχουν οι κατάλληλες δικλείδες ασφαλείας εδώ. Τώρα αυτή η προθεσμία της μίας ώρας ε, μου φαίνεται μη ρεαλιστική, εντελώ συμβολική. Θα πρέπει να βρούμε μια πιο λογική λύση εδώ. Πόσο μάλλον που είμαι και η συγκήτρια για ένα άλλο θέμα που αφορά τη συνεργασία μεταξύ των FIU όπου τα κράτη-μέλη και ιδιαίτερα το δικό μου κράτο είναι κατά οποιασδήποτε προθεσμία και οποιαδήποτε υποχρέωση ανταλλαγή πληροφοριών που θα μπορούσε να είναι χρήσιμη σε μια έρευνα για να εντοπίσουμε και να συλλάβουμε τρομοκράτες. Αυτό το κείμενο λοιπόν ε, είναι εξίσου σημαντικό με το άλλο και βλέπουμε εδώ ότι ακολουθούνται δύο μέτρα και δύο σταθμά και υπάρχει έχουμε να κάνουμε με δύο μέτρα τα οποία δεν είναι συμβατά μεταξύ τους. Λαμβάνω υπόψη λοιπόν όλα αυτά που διακυβεύονται ε, που σχετίζονται με τον κανονισμό αυτόν ελπίζω και πιστεύω ότι θα φτάσουμε σε μια δίκαιη και φιλόδοξη συμβαστική λύση για το κείμενο αυτό. Αναμένω με ανυπομονησία τη συνεργασία μας. Σας ευχαριστώ. Έχουμε καθυστερήσει αρκετά. Έχουμε και ένα σύντομο θέμα για τις ε, χρυσές ε, θεωρήσεις και μετά τις ε, ψηφοφορίες με την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων στις 4 και 4. Οπότε θα ζητήσω από τους άλλους συναδέλφους, τον κύριο Μπόνη και την κυρία Γκόμες, να είναι σύντομοι και να με συγχωρούν. Πρώτα ο κύριος Μπόνι. Ε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και να ευχαριστήσω τον κύριο Ντάλτον για το σχέδιο έκθεσης. Πολύ σημαντικό το θέμα. Και πρέπει να βρεθεί μια λίστα στο στόμα δυνατόν. Έχω κάποιες ερωτήσεις όμως. Μπορούμε να έχουμε σαφείς ε, ορισμούς ε, για το πως ο κανονισμός αυτός ε, σχετίζεται με την οδηγία του 2017. Έχω και εγώ κάποιες επιφυλάξεις επίσης για το χρονοδιάγραμμα της μίας ώρας. Γιατί, εντάξει, πρέπει να κινηθούμε γρήγορα, αλλά μία ώρα μπορεί να οδηγήσει σε λάθη. Ε, στο πώς θα αντιδράσουν οι αρχές. Δηλαδή, αυτό σημαίνει ότι οι πλατφόρμες θα αποφασίζουν το τι είναι τρομοκρατικό περιεχόμενο και αυτό πρέπει να το καθορίζει ο νόμος, όχι οι πλατφόρμες. Δεν θέλουμε να παραβιάσουμε εδώ πέρα τα πολιτικά δικαιώματα. Πρέπει επίσης ε, να υπάρχει ένας μηχανισμός προσφυγής κατά αυτών των αποφάσεων, εάν ε, γίνονται λάθη. Οι πολίτες ε, πρέπει να ξέρουν σε ποιον μπορούν να απευθυνθούν και να καθορίσουμε επίσης το τι θα γίνει με την ε, διατήρηση των ε, δεδομένων και να υπάρχει ένα κριτήριο διαφοροποίησης ε, των πληροφοριών από την πρόθεση της τρομοκρατίας. Ελπίζω λοιπόν να συνεχίσουμε σε αυτό το πνεύμα συνεργασίας. Ναι, Άννα, σύντομα παρακαλώ. Θα ήθελα να πω ότι δεν δέχομαι το ότι το κοινοβούλιο το καθυστερεί αυτό. Γιατί ποιος το καθυστερεί. Ποιος καθυστερεί την εφαρμογή ε, των πολύ κρίσιμων αυτών εργαλείων. Ε, τα κράτη-μέλη, το Συμβούλιο. Έγινε αναφορά στο θέμα της ε, συνεργασίας για την Μονάδα Οικονομικών Πληροφοριών που είχε ζητήσει η Europol και γενικά η εφαρμογή των οδηγιών για το ξέπλυμα χρήματος πραγματικά είναι αποκοστική ως προς τα αποτελέσματα που έχουν τα κράτη-μέλη. Συμφωνώ πλήρως με τους συναδέλφους που λένε ότι πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να τελειώσουμε εντός αυτής της θητείας. Πρέπει πραγματικά να γίνει αναφορά Ε, τα ζητήματα προστασίας δεδομένων αλλά το σημαντικότερο είναι η οδηγία ή η σχετική, γιατί δεν μπορούμε βεβαίως να έχουμε κάτι λιγότερο από την ελευθερία λόγου και συμφωνώ με τους συναδέλφους που αναφέρθηκαν ε, στο ότι πρέπει να υπάρχει δικαστικός έλεγχος ε, τελικά οι αρχές να κρίνουν το εάν θα πρέπει να αφαιρεθεί κάποιο περιεχόμενο. Σας ευχαριστώ. Κοιτάξτε, επειδή είναι σημαντικό το θέμα, ε, να σας παρακαλέσω να είστε λίγο σύντομοι. Γιατί έχουμε και άλλη μία παρουσίαση από την Κομισιόν. Οπότε δύο-τρία πράγματα ουσιαστικά και μετά θα επανέλθω στον εισηγητή. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ τον εισηγητή για το σχέδιο γνωμοδοτήσεως. Με τα χαράς βλέπουν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προχωράει Βάση της πρώτης συζητήσεως σήμερα πιστεύω ότι θα μας βοηθήσετε αυτή την πρόταση να την κάνουμε πιο ισορροπημένη και αυτό με κάνει ελπιδοφόρο ότι πράγματι μπορεί να υιοθετηθεί πριν το τέλος της θητείας. Αυτό είναι σημαντικότατο για μας. Υπάρχει τεράστια επιχειρησιακή ανάγκη για αυτή την νομοθεσία. Το τρομοκρατικό περιεχόμενο στο διαδίκτυο έχει παίξει το ρόλο σε πολλές τρομοκρατικές επιθέσεις σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και σίγουρα δεν είναι ένα μικρό πρόβλημα και ο όγκος τρομοκρατικού περιεχομένου στο διαδίκτυο είναι τεράστιος. Άρα χρειάζονται κάποια μέτρα τάχιστα. Να εστιαστώ επί τριών σημείων. Πρώτα απ' όλα επί του πεδίου εφαρμογής. Πολλοί από εσά το σχολιάσατε αυτό. Ευπρόσδεκτη κάθε προσπάθεια του Ευρωκοινοβουλίου να ρυθμιστεί καλύτερα το πεδίο εφαρμογής της, ε, του κανονισμού η πάροχη των διαφόρων υπηρεσιών νεφοϋπολογιστικών δεν ήταν στόχος μας. Μπορούμε να ρυθμίσουμε τις λεπτομέρειες του κειμένου. Μικρομεσαίες επιχειρήσεις όμως πρέπει να συμπεριληφθούν στο πεδίο εφαρμογής και σίγουρα δεν μπορούμε να τις εξαιρέσουμε από ιεσδήποτε υποχρεώσει στον τομέα για λόγους που απλώς θα τα συνδέονται με την επιχειρησιακή κατάσταση. Στην αρχή επικοινωθήκαμε των μεγάλων πλατφορμών, αλλά από όταν δραστηριοποιήθηκαν, τώρα το πρόβλημα διαδίδεται τάχιστα σε πολλές μικρομεσαίες πλατφόρμες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στον κόσμο. Αν τις αφήσουμε εκτός του πεδίου της προτάσεως, θα αποδυναμώσουμε την νομοθεσία και σε σημαντικό βαθμό. Πολλοί αναφέρθηκαν στον ορισμό του τρομοκρατικού περιεχομένου. Όλοι συμφωνούμε ότι πρέπει να βρούμε μια καλή ισορροπία ο ορισμός που προτείναμε εδράζεται επί της οδηγίας περί τρομοκρατίας και προσπαθεί να καλύψει το πιο επιβλαβές περιεχόμενο. Μιλάμε για υλικό που παρακινεί και ενθαρρύνει τρομοκρατικά αδικήματα, προωθεί τη δραστηριότητα τρομοκρατικής ομάδας ή δίνει οδηγίες σχετικά με την ε, πραγματοποίηση επιθέσεων. Και άλλοι περιορισμοί ε, όσον αφορά τον ορισμό είναι κάτι που να εξεταστεί προσεκτικότατα, διότι έτσι μπορεί θα είναι, μπορεί να δυσκολευτεί όλη η προσπάθεια να κατεβάσουμε περιεχόμενο τρομοκρατικό. Πολλοί αναφερθήκατε στον κανόνα της μιας ώρας. Θέλω να είμαι ακριβέστατος. Ο κανόνας της μιας ώρας ισχύει μόνο για νομικώς δεσμευτικά εντάλματα αφαίρεσης. Κάποιος δικαστής ή κάποια αρμόδια διοικητική αρχή έχει πιστεί ότι είναι παράνομο κάποιο περιεχόμενο και θα πρέπει να αφαιρεθεί. Η μόνη δράση που απαιτείται από εταιρείε σε αυτή την περίπτωση είναι να σταματήσουν την πρόσβαση στο περιεχόμενο. Δεν απαιτείται κάποια αξιολόγηση. Είναι δράσεις που μπορούν να αναλυφθούν τάχιστα. Ο κανόνας μιας ώρας βασίζεται επί στατιστικών στοιχείων που δείχνουν ότι η ζημιά που προκαλεί το τρομοκρατικό περιεχόμενο αυξάνεται δραματικά με κάθε ώρα στο διαδίκτυο. Τρομοκρατικές οργανώσεις έχουν δημιουργήσει συστήματα με αυτά εξασφαλίζουν το περιεχόμενό τους, μεταδίδεται τάχιστα σε διάφορες πλατφόρμες μετά την ανάρτηση. Όσο πιο γρήγορα κατέβει το περιεχόμενο, τόσο πιο αποτελεσματική είμαστε. Τελικό σχόλιο για τα ενεργά μέσα, μέτρα. Ακρογωνίος λίθος της προτάσεως είναι αυτός. Το σημαντικότερο κομμάτι πιθανότατα της προτάσεως και σχετίζεται απλούστατα με την κλίμακα του προβλήματος Μέχρι τώρα η μονάδα του διαδικτύου της Ευρωπόλ έχει καταγγείλει περίπου 63.000 τέτοιες αναρτήσεις τρομοκρατικές που έχει εντοπίσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Facebook από μόνο του, να είναι ένα παράδειγμα, διακόπτει ο Πρόεδρος, έχουμε παρουσίαση Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οπότε δεν έχουμε χρόνο, καταλαβαίνουν εκπρόσωπος της Κομισιόν, δύο προτάσεις μόνο. Το Facebook έχει αφαιρέσει 8,3 εκατομμύρια κείμενα από το περιεχόμενο σε τρει μήνες βάσει των δικών του εργαλείων. Οι εταιρείε ήδη ε, λαμβάνουν τα μέτρα, αλλά σήμερα δεν υπάρχει το κατάλληλο νομικό πλαίσιο, δεν υπάρχουν ε, ρήτρε διαφύλαξη, δεν υπάρχει προστασία. Και αυτό προσπαθεί να πετύχει εν λόγω πρόταση. Βασίζομαι στη βοήθειά σας, ούτω ώστε αυτές οι διατάξει να είναι ακόμα πιο καλά ισορροπημένε και να είναι ισχυρότερε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα. Σας ευχαριστώ. Κοιτάξτε, επειδή το επόμενο θέμα είναι η παρουσίαση της Κομισιόν για τις Χρυσέ Θεωρήσει και έχουμε 15 λεπτά τώρα, ε, δεν ξέρω τι να κάνω. Ναι, έτσι, σύντομα, σε παρακαλώ και θα δούμε τι θα κάνουμε. Θα ευχαριστώ, θα είμαι πολύ σύντομο, κύριε Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω όλους τους ε, συναδέλφους. Συμφωνώ με τι ε, περισσότερε παρεμβάσει Δεν απέχουμε πολύ. Προφανώς πρέπει να τα συζητήσουμε αυτά λεπτομερώς γιατί είναι ζητήματα δύσκολα. Ε, η πόρτα μου είναι πάντα ανοιχτή. Ε, νομίζω πρέπει ακριβώς να μπορούμε να ταυτοποιούμε το επικίνδυνο περιεχόμενο, το επιβλαβές και να το διαχωρίζουμε από το μη επιβλαβές και να δούμε τις πιθανές υποχρεώσεις. Αυτά θα είναι μια μεγάλη πρόκληση. Ε, για τα στατιστικά στοιχεία του Facebook πραγματικά κατέβασε εκατομμύρια αναρτήσεις χωρίς αυτή την ομοθεσία. Ε, πολλά πράγματα εθελοντικά. Ε, πρέπει να τα αναγνωρίσουμε και αυτό. Αλλά αναμένω βεβαίως την συνεργασία μαζί σας. Η πόρτα μου θα είναι άνοιχτη, όποτε θέλετε να συζητήσουμε. Και όπως είπα, αναμένω κάποια θετικά αποτελέσματα. Ναι, πράγματι το Facebook τα κατέβασε αυτά, αλλά δεν ξέρουμε τι, τι γίνεται. Δηλαδή, 8,3 εκατομμύρια από πόσα δεν ξέρουμε ακόμα και αν, ήταν κάποια, αν είχε κάποιο σοβαρό αντίκτυπο. Γιατί δεν, ε, δεν υπάρχει κάποιο πλαίσιο, είναι κάτι το εθελοντικό. Δεν ξέρουμε δηλαδή ποια είναι η συνολική κατάσταση και ε, βεβαίω και οι ίδιοι θα το παραδεχτούν. Αν και δεν ασκούμε κριτική βεβαίω για αυτό το οποίο έκαναν εθελοντικά. Είναι ένα τεράστιο θέμα το οποίο πρέπει να ε, ολοκληρωθεί μέχρι τις 15 του μηνός Οπότε σας ευχόμαστε καλή επιτυχία. Αλλά είναι τεράστια δουλειά. Το επόμενο θέμα είναι η παρουσίαση της Κομισιόν και ζητώ συγγνώμη από τους συναδέλφους της Κομισιόν γιατί έχουμε μόνο γύρω στα 20 λεπτά για να το παρουσιάσετε. την ε, έκθεση αυτή για την υπηκοότητα, για τους επενδυτές, ε, τις λεγόμενες χρυσές θεωρήσεις. Υπάρχει το έγγραφο το οποίο έχετε δει και ε, δεν ξέρω, μπορείτε να μας τα παρουσιάσετε σε τόσο σύντομο χρόνο. Εντάξει. Λοιπόν, αν μπορείτε να κάνετε μία παρουσίαση και ζητώ συγγνώμη από τους βουλευτές και ε, Άννα βεβαίως είναι το δικό σου το θέμα, εσύ θα μιλήσεις. Ε, προφανώς οι άλλοι βουλευτές τώρα ίσως χρειαστεί να τους περιορίσω τον χρόνο γιατί η πρώτη ψηφοφορία ξεκινάει σε 15 λεπτά, εντάξει. Εσάς. Και τέταρτο ψηφίζουμε, εντάξει. Ωραία. Λοιπόν, κινηθείτε αναλόγως. Ωραία. Τον λόγο έχει η Κομισιόν λοιπόν. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και ευχαριστώ και την Επιτροπή σας που μας δίνει μια δεύτερη ευκαιρία να παρουσιάσουμε αυτήν την πολύ σημαντική έκθεση γιατί αντιλαμβάνομαι πως η Επίτροπος η κυρία Γιούροβα είχε συζητήσει το θέμα με τα μέλη της Επιτροπής την προηγούμενη εβδομάδα για να κάνω μια σύντομη παρουσίαση θα ξεκινήσω από το 2014. Να σου πω ότι η πρόταση ξεκίνησε από το Κοινοβούλιο. Το Κοινοβούλιο ζήτησε από την Κομισιόν να αξιολογήσει διάφορα εθνικά σχέδια υπηκοοτήτων. Η ΔΕ Κομισιόν συνέταξε μια έκθεση το 2017 ε, είχαμε υποσχεθεί να κάνουμε μια, ένα απολογισμό και να δώσουμε και κατευθύνσεις στα κράτη-μέλη. Πριν από 10 μέρες πράγματι δημοσιεύσαμε την ε, σχετική έκθεση αλλά και ακόμη περισσότερα γιατί αν ε, και είχαμε δεσμευτεί να μελετήσουμε όλα τα εθνικά αυτά συστήματα πήγαμε παραπέρα γιατί αξιολογήσαμε και όλα τα σχετικά συστήματα που αφορούσαν την χρυσή βίζα, δηλαδή την άδεια παραμονής, όχι μόνο ε, υπηκοότητα δηλαδή, αλλά και την άδεια παραμονής. Θα σας παρουσιάσω λοιπόν την έκθεση, έκθεση η οποία βασίζεται στην πρώτη ε, μελέτη που είχε γίνει από μια εξωτερική εταιρεία, την Μιλιέ, που είχε περάσει από το σχετικό δίκτυο επαφών, είχε, βοηθήσει, είχε μελετήσει όλα τα σχετικά συστήματα των κρατών μελών, είχε και επαφές. Τέλος, με βάση αυτές τις ε, πληροφορίες συντάξαμε ένα έγγραφο εργασίας ε, το οποίο μας ε, εστιάζεται σε τρία κράτη, Βουλγαρία, Κύπρο και Μάλτα και εδώ πέρα σημαντικό είναι να πούμε ότι η Βουλγαρία εντωμεταξύ κατήργησε το σύστημα και σε 20 κράτη-μέλη όσον αφορά την χρυσή βίζα. Βουλγαρία, Κύπρο, Τσεχία, Εστονία, Ελλάδα, Ισπανία, Γαλλία, Κροατία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λετωνία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Ολλανδία, Πολωνία, Ρουμανία, Σλοβακία, Ηνωμένο Βασίλειο. Τι περιέχεται λοιπόν στην ε, έκθεση. Όπως σας είπα, οι εκθέσεις ε, καλύπτουν και τις δύο πτυχές, και την επικότητα και την άδεια παραμονής ε, και τις πληροφορίες για όλα αυτά τα συστήματα. Δηλαδή πόσα χρήματα πρέπει να επενδυθούν, ποιε είναι οι απαιτήσει για άδεια παραμονή, ποιοι είναι οι έλεγχοι ασφαλεία που κάνουν τα κράτη-μέλη, πώ συνδέεται ο έλεγχο ξεπλήματο χρήματο και τα σχετικά. Όλα αυτά θα τα δείτε στο έγγραφο εργασία. Επιπλέον, η Κομισιόν ε, εστιάζει και στο νομικό κομμάτι την νομιμότητα και των δύο περιπτώσεων και δείχνει σε ποιο βαθμό υπάρχει κοινωτική αρμοδιότητα. Τα κύρια ευρήματα είναι ότι η απόφαση ενός ε, κράτους μέλους για την απόδοση υπηκότητας ε, μέσω επένδυσης αυτομάτως επηρεάζει την σχέση με τα άλλα κράτη-μέλη. Εν σε ένα κράτος μέλος αποφασίζει και επηρεάζονται όλα τα κράτη-μέλη με την ε, απόδοση υπηκότητας. Με την άδεια παραμονής είναι εξίσου δραματική κατάσταση γιατί η απόφαση ενός ε, κράτους μέλους να δώσει άδεια παραμονής επηρεάζει το άτομο αυτό το οποίο μετά μπορεί να ταξιδεύει ε, για 20 μέρες κάθε 180 μέρες στην περιοχή Σέγγεν και παραπέρα. Οπότε το κυριότερο έβριμα μας είναι ότι τα συστήματα αυτά επηρεάζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της. Δημοσιεύσαμε και τις ε, πληροφορίες για τα αδύνα, αδύναμα στοιχεία. Ε, υπάρχουν αντικειμενικά στοιχεία που δείχνουν ότι για τρία κράτη-μέλη όπου ισχύει αυτό το σύστημα δεν απαιτείται να υπάρχει αυτοπρόσωπη παρουσία και κατοικία και παρομοίως ε, για την βίζα ε, υπάρχει μια τυπική απέτηση κατοικίας στα κράτη-μέλη. Επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό να πούμε ότι ενώ οι ετούντες έχουν υπηκότητα δεν χρειάζεται να αποδείξουν ε, κανέναν δεσμό με καμία από τις τρεις ε, χώρες ε, που δίνουν υπηκότητα. Δεν υπάρχει ανάγκη να υπάρχει δεσμός. Για την άδεια παραμονής επίσης υπάρχουν κάποιες ανησυχίες γιατί τα συστήματα αυτά ίσως να επηρεάζουν ε, την οδηγία περί μακροχρόνιας παραμονής. Ε, λοιπόν, έχουμε εν ολίγη στο θέμα της ασφάλειας, γιατί δεν είμαστε πεπισμένοι ότι η ε, έλεγχη ασφαλείας που κάνουν τα κρατη είναι αρκετά ε, σοβαρή. Βλέπουμε τη δυνατότητα να παρισφρήσει το οργανωμένο έγκλημα και υπάρχει κίνδυνος διαφθοράς. Υπάρχει σοβαρή ανησυχία για ζητήματα ξεπλήματος χρήματος, γιατί αυτή τη στιγμή τα συστήματα αυτά δεν ε, συμμορφώνονται απαραίτητος με τη σχετική νομοθεσία και όσον αφορά την υπηκότητα και όσον αφορά τα, την άδεια παραγωγής. Γι' αυτό ακριβώς εμείς προτείνουμε στα κράτη-μέλη να διοχετεύονται οι επενδύσεις αυτές μέσω των αρμοδίων αρχών. Τρίτον, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος φόρο διαφυγής λόγω των πιθανών λαθών και παρεξηγήσεων. Και τέλος, υπάρχουν σοβαρέ κίνδυνοι όσον αφορά την διακυβέρνηση και την διαφάνεια γιατί δεν υπάρχουν πληροφορίες από τα κράτη-μέλη, δεν υπάρχουν πληροφορίες για τους ελέγχους ασφαλείας, δεν υπάρχουν μηχανισμοί συνεργασίας ε, μεταξύ των κρατών μελών, π.χ. Δεν υπάρχει διαφάνεια επίσης ε, όσον αφορά τους αριθμούς των αδειών, ε, τους αριθμούς των αιτήσεων, τους αριθμούς των απορρίψεων και του συνολικού ε, εισόδηματος και του συνολικού οικονομικού ωφέλους. Η μελέτη δείχνει ότι το όφελος επίσης ήταν αρκετά περιορισμένο και υπάρχουν και κάποιες αμφιβολίες για την πιθανή σύγκρουση συμφερόντων. Σας παρακαλώ όμως συντομεύετε. Να σας πω λοιπόν τι σκοπεύουμε να κάνουμε. Αν έχετε διαβάσει την έκθεση ξέρετε ότι σκοπεύουμε να συστήσουμε μια ομάδα ειδικών μεταξύ των κρατών μελών με στόχο να υπάρξει κοινή έλεγχη ασφαλείας μεταξύ των οποίων και η διαχείριση του κινδύνου και θα εξετάσουν ε, τη χρηστή διοίκηση και την διαφάνεια. Έχει συνεδρι... Σκοπεύουμε να συνεδριάσει τρεις φορές μέχρι το τέλος του έτους η ομάδα αυτή και να υπάρξει και η απαραίτητη συνέχεια όσον αφορά την συμμόρφωση των συστημάτων αυτών με το κοινοτικό δίκαιο. Ανέφερα την οδηγία περί μακροχρόνιας παραμονής, κανόνες Σέγγεν, οδηγία ξεπλήματος ε, χρήματος ε, και την μελλοντική πέμπτη οδηγία. Θέλουμε επίσης να κινηθούμε προληπτικά όσον αφορά τις αρμόδιες αρχές και να δούμε τα ζητήματα της φοροδιαφυγής στην στενή συνεργασία με τα κράτη-μέλη. Λοιπόν, σταματάω εδώ, λέγοντας πως η Κομισιόν έκανε αυτό που της ζητήθηκε και θα δείτε ότι η έκθεση μας είναι πολύ καλή. Ευχαριστώ. Λοιπόν, δύο μιλητέ μόνο, διότι έχουμε την ψηφοφορία στα 3 και 4 και θέλουμε να διακόψουμε αμέσω πριν. Η κυρία Γκόμε και η κυρία Ίντεβελ. Δύο μιλητέ μόνο, παρακαλώ. Άννα πρώτα. Ναι, θα ήθελα να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την έκθεση. Είναι σημαντική και περιγράφει μια κατάσταση πολύ χειρότερη από αυτή που φανταζόμουν. Πολύ χειρότερη. Και δεν είναι μόνο ο αριθμό των κρατών μελών που εφαρμόζουν αυτά τα προγράμματα είναι οι επιπτώσεις, τα συμπεράσματα της Κομισιόν, πέρα από το ηθικό ζήτημα που τα κράτη-μέλη διαυκολύνουν ε, την χορήγηση χρυσών θεωρήσεων ενώ δεν αφήνουν πρόσφυγες και μετανάστες να φτάσουν στο έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διαφθορά, η φοροδιαφυγή, το ξέπλυμα χρήματο, η μεγάλη κίνδυνη και βεβαίω η κίνδυνη ασφάλεια γενικότερα, γενικότερα, γενικότερη που ανέφερε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διότι είναι, αυτό είναι ένα πρόγραμμα για να μπορέσει το οργανωμένο έγκλημα να διδεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το έχουμε δει αυτό. Με το Panama Papers ε, έχουμε πολλά παραδείγματα. Το πιο πρόσφατα είναι με τους Ρώσους στη Φιλανδία. Με το διαβατήριο το μαλτέζικο με εκατομμύρια από τράπεζες εστονικές ε, από τη Συρία ενώ υπήρχαν κυρώσεις για πωλήσει χημικών όπλων στο καθεστώς του ε, του Άσαντ άνθρωποι οι οποίοι βρέθηκαν ξαφνικά με χρυσή θεώρηση στην Ουγγαρία ε, κανένας από τα κράτη-μέλη η, η βασική ε, δέουσα επιμέλεια που χρειάζεται στις περιπτώσεις αυτές στη χορήγηση αυτών των θεωρήσεων. Είναι πραγματικά εξοργιστικό. Δεν μπορεί αυτό το κοινοβούλιο απλά να ακούσει την έκθεση αυτή και να μην κάνει τίποτα. Σας ζητώ λοιπόν, Πρόεδρε, ε, να υπάρξει ένα ψήφισμα στην τελευταία ε, ολομέλεια του Απριλίου με σαφή συστάση για τα κράτη-μέλη, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και για το επόμενο κοινοβούλιο, διότι αυτό το θέμα ε, δεν μπορούμε να το προσπεράσουμε και ελπίζω η Κομισιόν να ξεκινήσει διαδικασίες επιπαραβάση για τα κράτη-μέλη που έχει αποδειχθεί ότι έχουν παραμελήσει πολύ βασικά στοιχεία της ασφαλείας μας και που έχουν ενισχύσει το ξέπλυμα χρήματος. Και ένα ερώτημα προς την Κομισιόν δεν αναμένω βέβαια απάντηση γιατί το θέμα του καθεστώτος κυρώσεων ε, ε, δεν αναφέρεται εδώ και τις καθεστώ των κυρώσεων. Η κυρία Ιντεβελτ, ναι, ακούστε, εγώ είμαι κάπως λιγότερο ικανοποιημένη από την ε, έκθεση της Κομισιόν. Είναι κάπως αδύναμο. Αφού η Κομισιόν φτάνει στο συμπέρασμα ότι αυτές οι χρυσές θεωρήσεις, τα χρυσά διαβατήρια και αυτά τα προγράμματα αποτελούν κίνδυνο για την ασφάλεια, δεν μπορεί η Κομισιόν να προτείνει απλά την δημιουργία μιας ομάδας εργασίας όταν μιλάμε για άλλες μορφές εγκληματικότητας, η Κομισιόν ε, δεν θα ήταν τόσο χαλαρή. Ε, εδώ βέβαια μιλάμε για εγκληματίες ε, που δεν είναι μικροεγκληματίες, έτσι. Είναι πλούσιοι άνθρωποι, εύρωστοι, που δίνουν πολλά χρήματα στα εθνικά ταμεία. και αυτό είναι διαφθορά. Η Κομισιόν λοιπόν θα πρέπει να σταματήσει να μιλά για αρμοδιότητες της Ένωσης, να προτείνει να καταργηθούν αυτά τα προγράμματα. Διότι εδώ μιλάμε για την πώληση ευρωπαϊκής ηθαγένειας. Μιλάμε και για κάτι το οποίο έχει πολύ μεγάλο αντίκτυπο και στη Σέγγεν και σε ζητήματα ασφάλειας των Ευρωπαίων πολιτών. Αυτά τα προγράμματα ε, ουσιαστικά είναι ανήθικα, είναι ένα κόκκινο χαλί για απατεώνες και το λιγότερο που θα μπορούσε να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι να προτείνει μια διαδικασία όπως και για οποιοδήποτε καθεστώς ε, ηθαγένειας ή διαμονής για, τα, για τους ετούντες άσυλο υπάρχουν κοινέ διαδικασίες, υπάρχουν ε, κοινά κριτήρια, προϋποθέσεις. Αυτό είναι το λιγότερο που θα έπρεπε να κάνει η Ευρωπαϊκή, Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχω κάποιες ερωτήσεις. Θα ήθελα η Κομισιόν να μας πει, να ολοκληρώνω Κλοντ, ποιοι είναι οι συμμετέχοντες στην ομάδα πυρογνωμόνων και ποια είναι η μέρουσα διάταξη. Και τα πρακτικά. Θα ήθελα επίσης να γνωρίζω γιατί η Κύπρος από ό,τι φαίνεται αποχώρησε από την πρώτη συνεδρίαση που έλαβε χώρα τον Οκτώβριο. Θα θέλαμε να ξέρουμε γιατί. Επίσης, πότε θα ξεκινήσει μια διαδικασία επί παραβάση κατά των κρατομελών που δεν ζητούν από τους κάτοχους να διαμένουν πραγματικά στην χώρα ή να έχουν κάποια σχέση με αυτή τη χώρα. Το πιο σημαντικό πάντως, Πρόεδρε, είναι να δημοσιοποιήσει η Κομισιόν τον αριθμό των συμμετεχόντων, τα πρακτικά και την μέσα διάταξη αυτών των συνεδριάσεων της ομάδας εμπειρογνωμόνων. Ευχαριστώ. Ναι, να ζητήσω συγγνώμη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ξέρω ότι δεν έχετε χρόνο να απαντήσετε σε όλα αυτά τα σημεία και ζητώ συγγνώμη γι' αυτό. Θα πρέπει να γίνει γραπτό. Να δοθεί γραπτό η απάντηση. Έγινε κάποιε προτάσει από του ομιλητέ. Ε, παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον το ζήτημα. Ε, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί το ζήτημα αυτό. Είναι λίγος ο χρόνος, θα το συζητήσουμε με τους συναδέλφους και με τους συντονιστές. Δεν ξέρω, ε, μπορείτε να απαντήσετε γραπτός. Είναι σημαντικό αυτό, γιατί τώρα να περάσουμε ψηφοφορία. Ε, συγγνώμη που έτσι κάπως περιόρισα τη συζήτηση του θέματος αυτού. Ευχαριστούμε και για τις απαντήσεις, για το ζήτημα αυτό των χρυσών θεωρήσεων και των χρυσών διαβατηρίων. Λοιπόν, σε ένα λεπτό θα ξεκινήσουμε την ψηφοφορία με την Επιτροπή Γιούρη, οπότε ετοιμάστε τις κάρτες σας.